υπογραμμίζω ότι ο εξτρεμισμός είναι κάτι απαράδεκτο για την κοινωνία μας στο σύνολό της. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ και σας ευχαριστώ όλους για τις σημαντικές σας παρεμβάσεις. Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στο συντάκτη της προφορικής ερώτησης, τον συνάδελφο Λόπες Αγγιγιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διατυπώσαμε αυτή την προφορική ερώτηση μετά από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11 Σεπτεμβρίου 2012 σε σχέση με τις παράνομες πτήσεις στη ΣΥΑ και τις παράνομες επίσης κρατήσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος. Γιατί θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στο προηγούμενο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό έχω την τιμή να θέσω αυτό το προφορικό ερώτημα Προ την Κομισιόν καταρχήν για να ξέρουμε αν υπήρξε πλήρης διερεύνηση των παραβιάσεων τη κοινοτική ε, νομοθεσία σε ό,τι αφορά το άσυλο και την δικαστική συνεργασία. Αν υπήρξαν μέτρα τα οποία ελήφθησαν για να αποτραπεί ενδεχόμενη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ε, ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά και για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο των υπηρεσιών πληροφοριών τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια των επιτροπών της Επιτροπής Έρευνας που έχει δημιουργηθεί μέσα στην ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για τις ε, δράσεις μαζικής παρακολούθησης. Δεν πρέπει να υπάρχουν μαύρες τρύπες στη κοινωνία μας. Πρέπει όμως να θέσουμε το ερώτημα αυτό και προς το Συμβούλιο για να ξέρουμε αν υπήρξε η σωστή συνεργασία μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί μας δόθηκαν κάποια πρακτικά τα οποία είχαν μακιγιαριστεί από το Συμβούλιο. Αν γνωρίζει το Συμβούλιο λοιπόν ποια είναι η πραγματικότητα στα κράτη-μέλη και αν υπάρχει μια μεγαλύτερη θέληση να γίνει σαφής ο ρόλος των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών και το κατά πόσο συνεργάστηκαν με την CIA για αυτές τις δράσεις Απαγωγή ατόμων και παρανόμης κράτησή του. Πρέπει να ξέρουμε ποιε είναι οι χώρε όπου έχουν λάβει η χώρα με πιο έντονο το χαρακτήρα τέτοιου είδου ενέργειε. Η Λιθουανία που είναι τώρα η Προεδρία τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια χώρα που θίγεται από αυτέ τι καταγγελίε, αλλά το ίδιο αναφέρεται και για χώρε όπω η Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώ τι συνέβη, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια διευκρίνηση τη δράση τη CIA και να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα αυτά. Και για να διαλύσουμε οποιαδήποτε εντύπωση ότι υπάρχει ατιμορρησία αυτών των ανθρώπων σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές. Είναι απόλυτα απαράδεκτο να μπορέσουν να λάβουν χώρο, χώρα όλες αυτές οι ενέργειες στο ευρωπαϊκό έδαφος. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ποιος τις έχει διαπράξει, πώς έχουν διαπραχθεί και με ποιο τρόπο μπορούμε να αποτρέψουμε την επανάληψή του στο μέλλον. Δεν φαίνεται ότι οι έρευνες έχουν καταλήξει σε τίποτα προς το παρόν. Γι' αυτό εμείς καταθέσαμε την προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν και επίσης έχουμε και ένα ψήφισμα το οποίο έχουμε για τη λήξη της συζήτησης και ζητούμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για να υπάρξει ένα στεναρό μήνυμα προς το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη που να τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει τις ευθύνες του και θα παρακολουθήσει το θέμα αυτό. Ο κύριος Μπροκ, ο οποίος επίσης είναι συντακτής της ερώτησης αυτής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, μετά τις 9 Σεπτεμβρίου, λάθος, μετά τις 11 Σεπτεμβρίου, λέει ο κύριος Μπροκ, έχουν γίνει πάρα πολλά, τα οποία έχουν διαταράξει τους ε, κανόνες ε, συνεργασίας ε, και του κράτους δικαίου. Πρέπει λοιπόν να καταστήσουμε σαφές ότι αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Επίσης πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι οφείλουμε να βρούμε κανόνες για το κράτος δικαίου, οι οποίοι όμως κανόνες παράλληλα θα καταπολεμούν και την τρομοκρατία. Πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ο εχθρός μας δεν είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν πρέπει να προκαλείται αυτή η εντύπωση στη συζητήση μας. Και επίσης πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι σε ένα κράτος δικαίου όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε πρέπει να συζητούνται και αυτά τα θέματα με κριτικό πνεύμα. Και τα λέω αυτά για να μην δημιουργηθεί ε, λάθος εικόνα για τη στάθμιση των εξελίξεων και γεγονότων. Ελπίζω λοιπόν ότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα μας βοηθήσουν ε, θα απαντήσουν στα ερωτήματά μας. Βέβαια πρέπει να πω ότι υπάρχουν κάποια δύσκολα θέματα. Ε, αυτό το δυνητικό, το could clarify, αυτό είναι σημαίνει ότι και για μας πολλά πράγματα δεν είναι σαφή. Άρα δηλαδή εκφράζονται κάποιες εικασίες, κάποιες παραδοχές. Δεν είμαστε πάντα σίγουροι για το τι ακριβώς ε, συμβαίνει. Ε, θέλω όμως ε, να το συνδέσω όλο αυτό με τη συζήτηση που τρέχει τώρα και αφορά την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας, την NSA των Ηνωμένων Πολιτειών. Να στηρίξω την κυρία Αντιπρόεδρο ότι όσον αφορά θέματα ε, ενημέρωσης των πολιτών παραδείγματος χάρη στις ε, Ενωμένες Πολιτείες πρέπει να προχωρήσουμε πιο πολύ αυτή είναι πλέον η ευκαιρία μας να στρέψουμε το βλέμμα προς τα εμπρός να προχωρήσουμε στην προστασία των δεδομένων σε θέματα κράτος δικαίου να αναζητήσουμε προς τα εμπρός επικοδομητικές λύσεις οι οποίες αργότερα θα βοηθήσουν ώστε να μην επαναληφθούν καταστάσεις. Πρέπει να βρούμε κανόνες οι οποίοι δεν θα θέτουν το κράτος δικαίου στην υπηρεσία των αρχών ασφαλείας. Αυτό είναι λάθος. Και αυτούς τους συσχετισμούς πρέπει να τους ξεκαθαρίσουμε. Γι' αυτό πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία πλαίσιο για τα δεδομένα. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι απόλυτα σημαντικά. Πρέπει να γίνουν αυτοί οι συσχετισμοί, παραλαμβάνω, για το μέλλον. Να αναζητούμε πιο ισχυρές νομικές λύσεις. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ είμαι συντάκτης, ε, συνσυντάκτης ε, της ερώτησης, όχι του ψηφίσματος. Ε, θέλω να πω καθαρά, ηρωνικά και μην με παρεξηγήσετε, ότι η δική μου χώρα έχει προχωρήσει γιατί τουλάχιστον έχει απαντήσει σε κάποιες επιστολές. Εκ μέρους του Συμβουλίου, ο Υπουργός Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Σας είμαι ευγνώμων για τη δυνατότητα που μου δίνετε να απαντήσω στα διάφορα ερωτήματα που τίθενται στην προφορική ερώτηση που υπευλήθη από την Επιτροπή σας, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλα τα θεσμικά μας όργανα. Η εθνική ασφάλεια παραμένει ευθύνη των κρατών μερών. Αυτά λέει η συνθήκη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν υπηρεσίες πληροφοριών των χωρών μελών και αυτές είναι εκτός αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Οργάνων οι έρευνες ε, μικαζόμενων ε, υποθέσεων από πλευράς της CIA είναι θέμα λοιπόν των χωρών μελών. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών. Είναι κάτι που δεν μπορεί να με το οποίο να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λέει η συνθήκη και ακριβώς γι' αυτό το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στο ψήφισμά σας, το οποίο εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2012. Απλώς δεν είναι δυνατόν να εκπονεί δηλώσεις το Συμβούλιο σχετικά με τις υπηρεσίες των χωρών μελών. Είναι εκτός αρμοδιότητάς του και γι' αυτό ακριβώς το Συμβούλιο δεν είχε ούτε και ακροάσεις με τους αρμόδιους για την ασφάλεια των χωρών μερών είναι ένα θέμα που διμερώς με τα κράτη-μέλη συζητιέται. Δεν είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου να προτείνει ρήτρε ασφαλείας ώστε να διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διαδικασίες πληροφοριών ή να βάζει όρια στις υπηρεσίες αυτές και στις δραστηριότητε τους. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα νομικό για το Συμβούλιο και για όλα τα θεσμικά όργανα. Γι' αυτό το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να αναλάβει πρωτοβουλία για τίποτα προκειμένου να δοθεί συνέχεια στο περσινό σας ψήφισμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το Συμβούλιο σιώπησε πολλές φορές, με πολλές ευκαιρίες, είπε ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να λαμβάνει η χώρα με σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως επίσης πρέπει να γίνεται βάση της νομοθεσίας για την προστασία προσφύγων, κρατούμενων κλπ. Και ενώ δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί αυτό δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Μπορούμε να πετύχουμε τη μάχη κατά της τρομοκρατίας εφόσον παραμείνουμε πιστοί στις βασικές μας αξίες. Οποιαδήποτε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου από υπηρεσίες, κυβερνήσεις και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας τελικά μπορεί να ενθαρρύνει ορισμένα μεμονωμένα άτομα προς την τρομοκρατία. Και όχι το αντίθετο. Τέτοιες πράξεις λοιπόν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποτέ σαν άλοθη κάτω από καμία περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διάλογο με τις Ηνωμένε Πολιτείες όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο διάλογος αυτός είναι μια ευκαιρία για να συζητάμε ζητήματα όπως για παράδειγμα η κράτηση, ανάκριση, μεταφορά υπόπτων. Επιτρέπει επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογραμμίσει τη σημασία που δίνει στην τήρηση του διεθνούς δικαίου για των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως για να είμαστε σαφείς, συγκεκριμένες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφοριών δεν καλύπτονται από το διάλογο αυτό. Το Κοινοβούλιο έχει στη διάθεσή του πρακτικά τέτοιων συναντήσεων, όχι όμως πλήρη, συνοπτικά, διότι είναι θέμα απορρίτου. Διπλωματικές ανταλλαγές όπως αυτή έχουν μεγάλη αξία εφόσον οι συμμετέχοντες μπορούν ελεύθερα να εκφραστούν. Για τέτοια ευαίσθητα ζητήματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διπλωματία είναι πιο αποτελεσματική από ότι αν ανοιχτά τα πρακτικά κυκλοφορούν. Δεν πιστεύουμε ότι έχουμε παραβεί οποιαδήποτε αρχή όσον αφορά τα πρακτικά. Νομίζω ότι έχουμε τηρήσει τους κανόνες και τις πρακτικές. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, ο καθένας μας λειτουργεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που πρέπει να τηρούμε. Εκεί όπου μπορούμε να έχουμε πρόοδο ή να αναλάβουμε κάποια μέτρα, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Όπως στην περίπτωση του διαλόγου που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν θέλουμε να τηρήσουμε τις αρχές αυτές που σας ανέφερα πριν και να γίνονται σεβαστές από όλους, ο καλύτερος τρόπος είναι μέσω διπλωματίας και μέσω διακριτικού διαλόγου. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να είμαστε αποτελεσματικοί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ και τώρα το λόγο έχει αντιπρόεδρος η κυρία Ρέντινγκ οι πρακτικές που αναφέρονται ως παράνομες απαγωγές αποτελούν παραβίαση πολλών θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περιλαμβάνουν την παράνομη σύλληψη, την κράτηση και πολύ συχνά τα βασανιστήρια και την κακομεταχείριση. Και νομίζω έχουμε υπογραμμίσει επανειλημμένα ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιου είδους πρακτικές και ε, αυτό επιβεβαιώθηκε και από την Προεδρία του Συμβουλίου. Η Προεδρία του Συμβουλίου όμως υπογράμμισε και ένα άλλο γεγονός ε, θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας ε, είναι εκτός ε, των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη δεν δίνει αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνει έρευνες σε τέτοιου είδους θέματα. Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή ανέκαθεν υπογράμμιζε ότι εναπόκειται στα κράτη-μέλη να προβούν σε αντικειμενικές και αμερόληπτες έρευνες για να εξακριβώσουν την αλήθεια. Αυτό είναι μια υποχρέωση που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να διαπιστωθούν οι ευθύνε και για να μπορούν τα χρήματα να διεκδικήσουν και να αποκτήσουν αποζημίωση για τη ζημιά που έχουν υποστεί. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, διαβουλεύεται και πάλι για την παραβίαση διατάξεων από εκείνα τα κράτη, τα οποία από ό,τι φαίνεται συνεργάστηκαν στο πλαίσιο ενός προγράμματος της CIA. Αυτά αφορούν κυρίως την δικαστική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, ε, θα σας παρουσιάσω τα γεγονότα. Όταν Υπήρχε αυτό το πρόγραμμα και εφαρμόζεται από το 2001 μέχρι το 2003. Τότε δεν υπήρχαν ε, κοινοτικέ διατάξει που να αφορούν στη δικαστική συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Μόνο τον Οκτώβρη του 2009 το Συμβούλιο ενέκρινε μία απόφαση που έλεγε ότι θα πρέπει να συναυθούν δύο συμφωνίε με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Η μία θα αφορά την ε, ε, αμοιβαία, την αμφίδρομη δικαστική αρρωγή και το άλλο τις παράνομες απαγωγές. Και τα δύο τέθηκαν ε, σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2010 και οι δύο αυτές συμφωνίες ορίζουν το νομικό πλαίσιο συνεργασίας για ποινικά αδικήματα, πλαίσιο συνεργασίας με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να προβώ σε σαφή διαχωρισμό ανάμεσα σε δύο γεγονότα. Καταρχήν, στην υποχρέωση να αποκαλύψουμε την αλήθεια αυτό εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να συντονίζει άμεσα ούτε να διευκολύνει τις εθνικές έρευνες σε τέτοιου είδους θέματα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να ε, συγκαλεί επιτροπές ε, ή να ορίζει δικαστές. Το Συμβούλιο βέβαια είναι σήμερα παρόν στη συζητήση μας και το Συμβούλιο έχει ήδη πει με απόλυτη σαφήνεια ποιες είναι οι δικές του ευθύνες πάνω σε αυτό το θέμα. Δεύτερο τώρα στοιχείο. Πρέπει να αποφύγουμε τις ε, επικαλύψεις, ε, την επανάληψη γεγονότων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, πρέπει πάντα να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μία βασική αλληγή στο νομικό πλαίσιο από τότε που προέκυψε το πρώτο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η θέση σε ισχύ της ε, Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ για τις παράνομες κρατήσεις. Εδώ ε, πρόκειται για την εφαρμογή του νόμου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει ότι αυτό το εργαλείο, όπως και άλλα πολλά άλλα σημαντικά ε, κατά της τρομοκρατίας θα εφαρμόζονται με έναν τρόπο απόλυτα συμβατό με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, πάνω λοιπόν σε αυτή τη βάση η Επίτροπος κυρία Μάλστρομ και οι υποφαινόμενοι στις 5 Μαρτίου του 2013 έστειλαν μια επιστολή στους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης όλων των κρατών μελών και υπογράμμισαν το πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και να υπενθυμιστεί ότι τα εργαλεία αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται με έναν τρόπο απόλυτα συμβατό με το χάρτη. Μόνο έξι κράτη απάντησαν. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, υπενθύμησαν για άλλη μια φορά το θέμα στα υπόλοιπα κράτη-μέλη στις αρχές Απριλίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ζήτησε και πάλι απαντήσεις και είπε ότι και αυτή θα απαντήσει γιατί δεν θέλουμε να παραμελήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα ε, για τη δικαστική ε, αρρωγή σε ποινικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Και τώρα ακολουθούν οι ομιλητέ εξ των πολιτικών ομάδων με πρώτον για δύο λεπτά τον κύριο Κουέλιου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Αντιπρόεδρε Ρέντιν, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, Το σκοπός δεν μπορεί να δικαιολογεί τα μέσα. Γι' αυτό εμεί καταδικάζουμε στεναρά τι. Ε, ε, καταχρηστικές και παράνομες ενεργείες κατά της τρομοκρατίας μεταξύ των οποίων τις έκτακτες μεταγωγές, την ε, ε, απαγωγή, την κράτηση χωρίς δικαστική απόφαση και τις εξαφανίσεις. Ζητούμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν, να μα δώσουν πλήρε πληροφορίε για τη συνεργασία του με τις Αμερικανικές αρχές. Θέλουμε να υπάρξει πολιτική παρακολούθηση του θέματο αυτού και έλεγχο των κινήσεων που έλαβαν χώροι και να υπάρξει έλεγχο όπω ζητήσαμε στην Ολομέλεια. Δυστυχώ, ορισμένα κράτη-μέλη δεν δέχτηκαν να ελέγξουν την συμμετοχή των υπηρεσιών πληροφοριών στο πρόγραμμα τη ε, ΣΥΑ. Είναι γεγονό ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα για αντικειμενικέ και ανεξάρτητε ε, έρευνε που θα καταδείξει την ευθύνη για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από διάφορες αρχές και που θα επιτρέψει την αποζημίωση και την επανόρθωση του κακού που έγινε στα θύματα και επίση την βεβαίωση ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί αυτό το γεγονό. Θεωρούμε ότι οι έρευνε που έχουν γίνει από τα κατημέρια θα πρέπει να βασίζονται σε, σε στεναρέ δικαστικέ αποδείξει βάσει των εθνικών δικαιακών συστημάτων και την ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει το Συμβούλιο να κάνει μια προσπάθεια για να ξεκαθαρίσει την εικόνα του σε σχέση με τα θέματα αυτά. Το απαιτεί το Κοινοβούλιο και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καταδεχτεί ποια κράτη-μέλη είχαν ευθύνε στα θέματα αυτά και να ε, εγγυηθεί ότι δεν θα ξαναψευστεί ενώπιον του Κοινοβουλίου όπως έχει στο παρελθόν πρέπει να εκφράσει την δέσμευσή του για την αξία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Και πρέπει να γίνει σαφές ότι η άποψή μου και των ε, μελών του κόμματός μου για διάφορα στοιχεία του ψηφίσματος έχουν να κάνουν με σημεία του κειμένου και όχι με το γενικό ε, αποτέλεσμα που θέλει να επιτύχει το ψήφισμα και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Φλότρου για το έργο που έχει φέρει σε πέρα από την Επιτροπή Ελευθεριών. Η κυρία Φαγιών έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε πριν από ένα χρόνο. Εγκρίναμε ένα ψήφισμα και ζητήσαμε μέσω αυτού να υπάρξει μια απάντηση για τις καταγγελόμενες μεταγωγές κρατουμένων στις νομές από τις ΗΠΑ και τη CIA. Η αλήθεια ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί. Ούτε μία χώρα και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο έχουν ακούσει τις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αποκάλυψη της αλήθειας. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτές τις εσχρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις χειρότερες αυτές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι κυβερνήσεις δεν θέλουν να συνεργαστούν, δεν υπάρχουν ανεξάρτητες έρευνες, αλλά αναδύονται συνέχεια καινούργια στοιχεία. Εδώ και πολύ καιρό έχουμε προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να κουκουλώσει τα σφάλματά της και τις ευθύνε της. Αλλά βλέπουμε να γίνονται συνέχεια τέτοια σφάλματα. Είδαμε την τραγωδία έξω από τις ακτές της Λαμπεδούσα που οδήγησε στο θάνατο πάνω πάνω από 300 προσφύγων από τη Συρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι το πιο σύγχρονο τμήμα του κόσμου. Όταν έχουμε όμως την τεράστια αυτή άγνοια, όταν επιτρέπουμε τόσο σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χάνουμε κάθε αξιοπιστία μεταξύ των πολιτών μας. Πώς μπορούμε μετά να ζητούμε από άλλους να φέρονται διαφορετικά. Πόσοι άνθρωποι πρέπει να πεθάνουν, πόσες ζωές πρέπει να χαθούν προτού συνειδητοποιήσουμε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι και πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε. της. Σήμερα, μετά από ένα χρόνο, εξακολουθούμε να μιλάμε για αυτές τις έκτακτες μεταγωγές, για την παραβίαση της κυριαρχικότητας των κρατών μελών, για την παραβίαση δικαιωμάτων και ελευθεριών που έχουν θεμελιώδη χαρακτήρα. Και εδώ πρέπει να αναφέρουμε και την παράνομη κράτηση, την κακομεταχείριση, την παραβίαση της αρχής μη επαναπρόθεσης και τις εξαφανίσεις ακόμα κρατουμένων. Όλα αυτά λοιπόν επαναλαμβάνονται και αυτά δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και τις CIA σε αυτά τα μυστικά προγράμματα. Ζητούμε λοιπόν από τη Λιθουανία να φέρει τη συζήτηση για τις ευρωπαϊκές ευθύνες στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού των αρμοδίων υπουργών στο, Ευρωπαϊκό, στο Συμβούλιο. Μας ε, απογοητεύει το γεγονός ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν απαντήσει καν στις επιστολές της Κομισιόν σε σχέση με τα προγράμματα αυτά. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων γεγονότων. Δυστυχώς βλέπουμε όλο και περισσότερες νέες σκανδαλώδεις ενέργειες, παρακολούθηση τηλεφώνων, φυλακίσεις κτλ. Δεν έχουμε λοιπόν καμία απάντηση στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από ένα χρόνο για τι καταγγελόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ευρωπαϊκό Έδαφο. Περιμένω λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι και κυρία Επίτροπε ότι αύριο θα υπάρξει πλήρης υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για, την, για το ψήφισμά μα, γιατί πρέπει να αναλάβουμε και εμεί τι ευθύνε μα σε σχέση με τη συνειδητοποίηση αυτών των παραβιάσεων. Υπάρχει μια πλεκάτα για σας κυρία Φαγιόν. Είσαστε έτοιμοι να απαντήσετε. Κύριε Λίσεκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε. Κυρία Φαγιόν, θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα. Σας ε, εκτιμώ ιδιαίτερα. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω αν έχετε διαβάσει τον τίτλο της σημερινής συζήτησης. Καταγελόμενες παράνομες μεταγωγές και κρατήσεις. Δεν υπάρχει κάποια έρευνα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος που να έχει υπερατωθεί. Οι έρευνες και <clears throat> οι διερευνήσεις είναι ακόμα εν εξελίξη. Μήπως, κυρία Φαγιόν, θα ήταν πιο λογικό να μιλήσετε για καταγγελόμενες μεταγωγές και υπο, υποψίες ε, παράνομης κράτης όσο δεν έχουν αποδειχθεί όλα αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Λίζε, για το ερώτημά σας. Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημά σας. Συμφωνώ μαζί σας ότι ο τίτλος του ψηφίσματος είναι «Καταγγελόμενες κρατήσεις και μεταγωγές». Στην πράξη όμως κάθε μέρα, η πραγματικότητα είναι ότι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα διαβάζουμε στα μέσα ενημέρωσης για νέες υποθέσεις οι οποίες έχονται στο φως. Είναι γεγονός ότι κανένα θεσμό, καμία κυβέρνηση δεν έχει ε, απαντήσει στις εκκλήσεις μας πριν από ένα χρόνο. Έχουν σταματήσει πολλές έρευνες, πολλές έρευνες δεν έχουν προχωρήσει ποτέ στη Λουθουανία Ισχύει αυτό μεταξύ άλλων. Επομένως κανείς δεν έχει αποκαλύψει πλήρως την αλήθεια και είναι μια ευκαιρία για μας να δείξουμε πόσο σοβαρές ήταν αυτές οι παραβιάσεις. <clears throat> κυρία Λάτφορτ έχει το λόγο. Το ψήφισμα αυτό δύο πράγματα κάνει. Το ένα είναι ότι επαναλαμβάνει την ίδια κριτική όσον αφορά το πρόγραμμα παράτυπων παραδόσεων ε, υπόπτων που οδηγούνται σε βασανισμούς και την συνενοχή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από δέκα χρόνια, κλείσαμε τον προηγούμενο μήνα, οργανώσαμε την πρώτη ακρόαση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Γουαντάναμο. Η νομική σκέψη οδήγησε σε στραβό Προηγουμένως όμως θέλω να επικεντρωθώ στο δεύτερο στοιχείο του ψηφίσματος που ζητάει λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο και από τη δικιά μου χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο και η Επιτροπή να βοηθήσουν ελέγχοντας και στηρίζοντας την άσκηση λογοδοσίας από τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν είναι εκτός αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συμβουλίου, έχω να πω εγώ στο Συμβούλιο, τότε γιατί έχουμε τέτοιες ε, ρήτρε ή τη Χάρτα Θεμελιωδών ε, Δικαιωμάτων. Τι νόημα έχουν οι δηλώσεις που κάνουμε όσον αφορά τις αντιτρομοκρατικές δράσεις που λέμε ότι πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν δεν δίνεται συνέχεια σε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο. Ενώ υπάρχουν τόσες πολλές αποδείξεις. Δεν πρέπει πια να αυτό το «Οικαζόμενες» να το διαγράψουμε από τον τίτλο διότι έχει υπάρξει παραβίαση αυτών των κανόνων και του διεθνούς δικαίου. Και έρχομαι τώρα πάλι στο διεθνές νομικό πλαίσιο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε προσπαθούν στα πλαίσια της μάχης κατά της τρομοκρατίας να παρακάμψουν τους νόμους. Έχει αλλάξει η ορολογία βέβαια. Ο Ομπάμα δεν μιλάει για τον πόλεμο όπως μιλούσαν οι προκάτοχοί του. Όμως οι Ηνωμένε Πολιτείε είδαν ότι έγινε με την επίθεση στην ε, Λιβύη την προηγούμενη εβδομάδα. Και το Γουαντάναμο εξακολουθεί να είναι ανοιχτό παρά το όσα είχαν υποθεί νωρίτερα και παρά το γεγονός ότι πάρα πολλοί δεν έχουν δικαστεί ακόμα. Το Συμβούλιο λοιπόν θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να ηγηθεί στην διερεύνηση της αλήθειας. Ως αντιπρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας του Πακού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, θέλω ό,τι καλύτερο από τις ΗΠΑ. Αλλά όταν το βαγόνι βγει από τη γραμμή, δεν το τραβάς για να βγει ακόμα περισσότερο, προσπαθείς να το βάλεις πίσω στις ράγες. Και δεν είναι αυτό που κάνει το Συμβούλιο σήμερα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Φλότρ τώρα για δύο λεπτά. Παρακαλώ κύριε Φλότρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως υπενθυμίστηκε εδώ και ένα χρόνο έχουμε μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από μια μακροσκελή και πάρα πολύ ενδελεχή που έγινε <clears throat> με επικεφαλή στον κύριο Κουέλιο από την Ερευνητική Επιτροπή για τις ε, έκτακτες αυτές παραδόσεις. Ήταν μια έκθεση που εγκρίθηκε με μια ευρύτατη πλειοψηφία και Ελπίζω ότι αυτή η συνένεση για τη δικαιοσύνη και την αλήθεια θα υπάρχει και πάλι αύριο όταν ψηφιστεί το σημερινό ψήφισμα. Το τωρινό μας ψήφισμα ενημερώνει το προηγούμενο σε σχέση με τις ενέργειες αυτές οι οποίες έχουν λάβει η χώρα και θα ήθελα να πω στον Πολωνό συνάδελφό μας ότι εδώ και ένα χρόνο υπήρξε η απόφαση του ΕΔΑΔ σε σχέση με τη δράση της Μακεδονίας σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εφέτος η Φιλανδία ανακοίνωσε μέσα του διαμεσολαβητή της μια έρευνα που έγινε και τόνισε ότι υπήρξαν καταδίκες για υπαλλήλου τη CIA και των Ιταλικών μυστικών υπηρεσιών. Όλα αυτά είναι έρευνες οι οποίες έχουν επερατωθεί, Αλλά έχουμε και νέα θύματα τα οποία έγιναν γνωστά και ζητείται η δικαιοσύνη στη Λιθουανία για αυτά τα θύματα. Αυτά ήταν πέρσι και επίσης το ίδιο είναι και για την Πολωνία ένα θύμα που ζητά να αναγνωριστεί το γεγονός ότι ήταν θύμα τέτοιων παράνομων ενεργειών. Κάθε μέρα λοιπόν έχουμε και νέα στοιχεία τα που έρχονται στο φως. Θα ήταν πραγματικά απόλυτα μάταιο τα κράτη-μέλη να θάβουν το κεφάλι του στόχο στην άμμο ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα ξεχαστούν όλα αυτά και δεν θα θελήσει κανείς ποτέ να ξέρει την αλήθεια. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται για να μπορέσουν να αποκαλύψουν την αλήθεια. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Προεδρία του Συμβουλίου που εκπροσωπείτε εσείς είσαστε Λιθουανός. Η χώρα σας πάντα είπε ότι θα κάνει μια έρευνα, ότι ήταν διατεθειμένη να κάνει κάτι τέτοιο εάν ερχόντουσαν στο φως νέα πραγματικά στοιχεία. Αυτά τα νέα στοιχεία υπάρχουν και σας παρακαλώ να μπορέσετε να, αναλάβετε τις ευθύνες σας για να δημιουργήσετε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο υποστήριξης αυτών των ερευνών στα κράτη-μέλη, ώστε επιτέλους οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν την εγγύηση ότι οι πολιτικές οι οποίες γίνονται προς όφελος της ασφάλειάς τους γίνονται μέσα στα πλαίσια της στήριξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο κύριος Κίρκοφ έχει το λόγο. 3,5 λεπτά εκ μέρους των ε, συντηρητών. Οι κατηγορίε οι αιτιάσεις ε, από τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να αγνοούνται. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ε, προσήκουσα σοβαρότητα. Η απάνθρωπη συμπεριφορά ποτέ δεν μπορεί να είναι ένα εργαλείο ε, το οποίο να, στο οποίο βασίζεται μια υγιής κοινωνία. Η δική μας η χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, είναι μια χώρα που εμπλέκεται σε αυτές τις αιτιάσεις, αλλά είναι μια χώρα με μακρά παράδοση ελευθερίας και κράτους δικαίου. Χαιρετίζω λοιπόν την ευκαιρία για αυτές τις ε, έρευνες για να αποκατασταθεί η φήμη μας που αυτή τη στιγμή έχει αμαυρωθεί. Βέβαια οι έρευνες πρέπει να γίνουν από μια πεπατημένη καθιερωμένη διαδικασία, απόλυτα ανεξάρτητη δικαστική αρχή ε, δεν πιστεύω όμως ότι το κοινοβούλιο αυτό είναι σε θέση να εκφράζει απόψεις για το πώς θα γίνονται οι έρευνες. Δυστυχώς εδώ οι αιτιάσεις πολλές φορές αντιμετωπίζονται ως ε, γεγονότα και οι συστάσεις αντιμετωπίζονται ως καταδίκες. Πρέπει να σταματήσει λοιπόν αυτό αν θέλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει σημαντικότερο ρόλο ε, Διερωτώ με όμως ε, γιατί, πώς είναι δυνατόν να αναλάβει αυτό το ρόλο με αξιόπιστο τρόπο. Δεν έχω ιδέα πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά ούτε και άλλοι οι οποίοι εφαρμόζουν και επιθυμούν να υπάρχει αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη για αυτό το θέμα. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε κύριε Σεπάνεν. Η κυρία Βερζιά έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και ένα χρόνο είχαμε εγκρίνει ένα κείμενο για τις δράσεις της CIA στο ευρωπαϊκό έδαφος. Ήταν ένα σημαντικό σημαντικός κρίκος στη διαδικασία διερεύνησης των ευθυνών για τα προγράμματα ε, μεταγωγών της ε, και παράνομης κράτησης της CIA. Έχουμε εκθέσεις μεταξύ άλλων και του Συμβουλίου της Ευρώπης και μετά από όλα αυτά ήταν απαραίτητο για την εισηγήτρια να αναλάβει την ε, ενημέρωση αυτού του φακέλου. Και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Φλότρο για όλα αυτά. Οι περισσότερες συστάσεις μας όμως δεν έτυχαν συνέχεια και οι περισσότερες έρευνε, όσε ξεκίνησαν δεν, δεν προχώρησαν καθόλου. Δεν αντιμετώπισαν καν τις νέες πληροφορίες οι οποίες έρχονται στο φω συνέχεια. Αυτή η αδράνεια είναι σκανδαλώδη. Μερικοί θέλουν να γυρίσουν πίσω και να παραμείνουν μονάχα στο επίπεδο γενικών σχολείων. Στο ψήφισμα το οποίο θα υποβληθεί αύριο, εμεί θα ακολουθήσουμε την ίδια γραμμή όπως και πέρσι. Θα παραμείνουμε στα γεγονότα. Ο καθένα θα πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε του και όπω είπατε κύριε Επίτροπε θα πρέπει να υπάρχει επανόρθωση εναντί των θυμάτων. Ήταν απόλυτα απαράδεκτες αυτές οι ενέργειες ανεξάρτητα από τα κράτη τα οποία εμπλέκονται. Κύριε Υπουργέ, εμείς σε αυτό το κοινοβούλιο θεωρούμε ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών είναι κάτι που μας εμπλέκει όλους. Σταματήστε να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλο και τις αρμοδιότητές σας και να αρνείστε να απαντήσετε στα ερωτήματα. Ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας δεν πρέπει ποτέ να οδηγήσει στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε αλήθεια, χρειαζόμαστε δικαιοσύνη. Αν υπήρξαν οριστήματα θα πρέπει να αναγνωριστούν και να τιμωρηθούν για να μην μπορούν να ξαναγίνουν τέτοιε ενέργειε. Και είναι καιρό επιτέλου να αναγνωριστεί αυτό. Ευχαριστώ. Εκ ε, των ε, Σοσιαλδημοκρατών, ο ε, μάλλον των Πάτεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε τις παράνομες μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη από τη ΣΕΕ και αυτό είναι λάθος. Οι ύποπτοι για ποινικές, ε, ποινικά εγκλήματα έχουν δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Βεβαίως αυτή η προφορική ερώτηση δεν αφορά αυτό. Πρόκειται για το ότι ζητάμε από την Κομισιόν να εισάγει περισσότερα μέτρα για να μπορούμε να ελέγχουμε την κατάσταση. Βεβαίως ε, οι πολίτες μπορούν να διαβάσουν περισσότερα στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει τον ε, τίτλο Ασφαλή κόσμος, καλύτερος κόσμος, στο πλαίσιο του προγράμματος της Στοκχόλμης. Οι προτάσεις αυτές είναι άλλο ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση για να δημιουργήσουμε, να συστήσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται και τον έλεγχο των υπηρεσιών ασφαλείας ε, εκτός από την εξωτερική πολιτική για να ολοκληρώσει την εικόνα. Βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αυτή τη στιγμή την αρμοδιότητα να το πράξει αυτό και εμείς δεν θέλουμε ποτέ και να την αποκτήσει. Most Ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Παπα-Νικολάου. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάνοντας μια, σύντομη αναδρομή, ε, θα έλεγα ότι πέντε χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η συζήτηση στο Κοινοβούλιο μας, κάποιοι από εμά δεν ήμασταν ούτε ε, εκλεγμένοι ευρωβουλευτές εδώ, ε, τότε υπήρξε μια έκθεση η οποία με τα, στοιχεία που υπήρχαν τότε και τις εκατέρωθεν καταγγελίες ε, κατέληξε σε κάποιο κείμενο το οποίο δεν στηρίχθηκε από όλους διότι κάποιες κατηγορίες κάποιες δηλώσεις θεωρήθηκαν τότε ότι δεν ήταν ακριβείς ότι ε, ήταν πολιτικά υποκινούμενες. τα αναφέρω αυτά κάποια χρόνια μετά για να ξεκαθαρίσω από την πλευρά όλων μας νομίζω ότι όλοι είμαστε υπέρ της προστασίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό σε κάθε περίπτωση. Όλοι είμαστε κατά τη παράνομη κράτηση συνανθρώπων μα και πρέπει να σεβόμαστε του νόμου και τι συνθήκε. Και φυσικά κάθε παραβίαση τη Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα. Αυτά είναι ξεκάθαρα και γι' αυτό το λόγο για πρώτη φορά εγώ πέρυσι που γνώρισα το θέμα στη διάσταση του κοινοβουλίου μας ψήφισα την έκθεση φλότρ και πολύ ευχαρίστως ένα τέτοιο κείμενο θα το ξαναψήφιζα. ένα χρόνο μετά όμως χωρίς να έχουν προκύψει πολλά νέα δεδομένα βλέπουμε ένα ψήφισμα που έρχεται αύριο προς ψήφιση το οποίο περιλαμβάνει μέσα κατηγορίες οι οποίες είναι αναπόδεικτες και ονοματίζει συγκεκριμένα κράτη μέλη χωρίς να προκύπτουν συγκεκριμένα στοιχεία. δεν μπορούμε να κάνουμε αναφορές με όρους επικοινωνίας ή με όρους πληροφοριών μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. χρειάζεται διερεύνηση χρειάζεται εξακρίβωση χρειάζεται νομική διαδικασία όπως αυτή ορίζεται σε κάθε κράτος μέλος κλείνω λοιπόν και επαναλαμβάνω είμαστε υπέρ και ξεκάθαρα υπέρ του απόλυτου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. είμαι πολύ επιφυλακτικό όμω για ένα ψήφισμα αύριο που περιλαμβάνει ανακρίβειε και κατονομάζει ψευδό σε πολλέ περιπτώσει από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω ε, μεμονωμένα κράτη μέλη. ευχαριστώ πολύ. Eh, ευχαριστώ. Η κυρία δύο θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελένη Φλόθο για τη δουλειά που έκανε, μας οδήγησε αυτή την έκθεση. Βλέπουμε κυβερνήσει των κρατών μελών σε χώρε υποψήφιες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και οι αρμόντες εθνικές αρχές ε, δεν δίνουν καμία απόκριση στα αιτήματα που έχουμε καταβάλει για την εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία των ε, θυμάτων στα πλαίσια του προγράμματος ε, της CIA και τους φυλακισμένους που βρίσκονται σε μυστικές φυλακές CIA μεταξύ των οποίων και τον Κουαντάναμο. Έχουμε καταθέσει νέες αιτήσει διευκρινήσεων για 28 συγκεκριμένες περίπτωση ε, στην Πορτογαλική επικράτεια ε, ε, από το 2001 μέχρι το 2006. Τον Οκτώβριο του 2011 έστειλε επιστολή στην τότε Πορτογαλική κυβέρνηση, αλλά δεν έχω λάβει έκτοτε καμία απάντηση. Υπάρχουν αποφάσεις ευρωπαϊκών και εθνικών δικαστηρίων και εκθέσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων που επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών σε αυτή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα εγκλήματα που διεπράκτησαν, οι αρμόδιοι για αυτά τα προγράμματα έχουν ενθαρρύνει την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, στην πολιτική καταπολέμηση τη τρομοκρατία ε, τόσο στην ΕΕ όσο και στη ΣΥΠΑ, όπω βλέπουμε στο πρόγραμμα PRISME τη NSA, Παραδείγματο χάρη, ή στο Operation Socialist ε, τη Αντίστοιχη GCHQ του Ηνωμένου Βασιλείου και την περίπτωση Belgacom. Η τρομοκρατία αυτή δεν μπορεί να καταπολεμηθεί ούτως ή άλλως και κυρίως όχι με αυτά τα μέτρα. Οπότε η οργανωμένη εγκληματικότητα με αυτήν την ατιμορρησία μας οδηγεί σε κλοπή προσωπικών δεδομένων και κυριως οχι με αυτα τα μετρα οποτε η οργανωμενη εγκληματικοτητα με αυτην την ατιμορρησια μας οδηγει σε κλοπη προσωπικων δεδομενων και παραβια τη ιδιωτική ζωή. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι μυστικέ υπηρεσίες, ε, τον είπα και οι Ευρωπαίοι ομότιμοι τους, ε, κατηγορούν τους πολίτες ε, αποδίδοντας και ατομικές και ευθύνε, ευθύνες αδικαιολόγητα. Βλέπουμε ότι είναι μια πελώρια ανοησία η απάντηση που μας δίνει το Συμβουλίο. Θα ήθελα λοιπόν να ε, ζητήσω να ξεκαθαριστεί η υπόθεση, να δούμε τις υποθέσεις ε, όπως εξελίσσονται τώρα στο Αμερικανικό Κογκρέσο, να ασκηθούν οι εθνικές αρμοδιότητες αλλά και οι ευρωπαϊκές αρμοδιότητες ε, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και δεν ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας και διαπραγματευόμαστε μια διατλαντική συμφωνία. Αυτή τη στιγμή ε, εξετάζεται η αναβολή των συμφωνιών PNR και SWIFT και διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λίσεκ θέλει να θέσει μία ερώτηση προς εσάς. Είστε έτοιμοι να απαντήσετε. Θα έχετε και λίγο χρόνο εξτρά. Κύριε Λίσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ καλή δουλειά κάνετε και την εκτιμώ. Χρησιμοποιείτε ωστόσο έναν όρο στην παρέμβασή σας που είναι συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών και NSA χαρακτηρίζοντάς τες ως εγκληματικού χαρακτήρα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό αφορά, στηρίζεται σε διεθνείς ή διμερείς συμφωνίες. Τι το ποινικό εγκληματικό έχει κάτι τέτοιο. Το ότι υπεξαιρούνται ε, στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών. Οτιδήποτε είναι κατά του νόμου ή ερμηνεύει ευρέως υφιστάμενες ε, ε, συμφωνίες και παραβιάζει με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματα των πολιτών δεν είναι σωστός τρόπος διεξαγωγής της μάχης κατά της δημοκρατίας. Ίσα ίσα που βοηθά τους, χρησιμοποιείται από τους τρομοκράτες γιατί ε, εντείνει τις υποψίες μεταξύ των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πιωτρόφσκι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στις προφορικές ερωτήσεις σήμερα και στο ψήφισμα για τις ε, εικαζόμενες ε, φυλακές της CIA στην Ευρώπη, το Κοινοβούλιο προσπαθεί να διαφυλάξει τα δικαιώματα του ανθρώπου. Οι μυστικές υπηρεσίε δεν έχουν θεωρητικά δικαίωμα σύλληψη. Το Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα, οποιαδήποτε αρμοδιότητα στον τομέα αυτό. Όλοι στο Κοινοβούλιο υποστηρίζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η ομάδα μου προτείνει μία ένα σύντομο και πολύ καλό ψήφισμα που αναφέρει ότι τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για να διαφυλάσσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να υποστηρίζονται. Εάν ωστόσο παρεμβαίνουμε στην λειτουργία των δομών αυτών, ρωτάω, θα θέτουμε συνεχώς ερωτήσεις και θα υιοθετούμε συνεχώς ε, ψηφίσματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Προτασίεβης τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αναμφίβολα οποιαδήποτε παραβίαση νόμων, οποιοδήποτε τέτοιες περιπτώσεις <clears throat> πρέπει να διευκρινιστούν, να διαλευκανθούν Πρέπει όλοι όσοι εμπλέκονται ε, σε τέτοιες υποθέσεις και εδώ στην Ευρώπη και από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Εκκρεμούν ορισμένες τέτοιες υποθέσεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Και αν βρούμε αποδεικτικά στοιχεία, ξέρετε ότι πολλές φορές μπορεί οι ποινές που θα επιβληθούν να είναι ιδιαίτερα βαριές. Είμαι πεπισμένος ότι εφόσον ε, καταδειχθεί ότι αυτές οι λεγόμενες ε, φυλακές ε, που αναφέρονται ότι υπήρχαν και στην Πολωνία υπάρχουν, τότε θα πρέπει να υπάρξουν εναγκαίες ποινές. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω μιας ανεξάρτητης έρευνας, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει στην Πολωνία και είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει κάθε καλή θέληση να διαλευκανθούν αυτοί οι ισχυρισμοί και βέβαια πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν είναι εύκολες αυτές οι περιπτώσεις Υπάρχουν ε, διαφορετικού τύπου προβλήματα για να διευκανθούν αυτές οι υποθέσεις. Και τα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών, όπως αναφέρει το ψήφισμα, ε, είναι αμφίβολο εάν μπορούν να συνελέσουν με αυτόν τον τρόπο, να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου είπε σωστά ότι τα θέματα αυτά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και αν δεν αναφερθούμε στα δικαστικά συστήματα στις εισαγγελίες φοβάμαι ότι δεν θα ε, μπορέσουμε να υποστηρίξουμε το ψήφισμα αυτό. Ε, κύριε Προτασίεβιτς, ε, έχει υπάρξει μια μπλε κάρτα. Θέλετε να απαντήσετε στην κυρία Φλότρα. Φλότρα, θα ήθελα να ζητήσω από τον συνάδελφό μας, εάν δεν νομίζει ότι για να υπάρχουν ανεξάρτητες έρευνες ε, προδιαγραφές που πρέπει να γίνουν σεβαστές και αν θεωρεί ότι παράγραφος 6 που ζητά από την Πολωνία να συνεχίσει τις έρευνές της με περισσότερη διαφάνεια και να συνεργαστεί ανεπιφύλακτα με τις αρμόδιες αρχές για να αντιμετωπιστούν οι διάφορες, ε, ε, οι χειρισμοί. Δεν θεωρεί ότι πρέπει να γίνει αυτό. Εμεί Εμείς είχαμε μετάσχει στις ακροάσεις που είχαν γίνει στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πριν λίγο καιρό και είχαμε την ευκαιρία να δούμε λεπτομεριακά την κατάσταση από χώρα σε χώρα. Για την Πολωνία και ανεξάρτητοι ακόμα παρατηρητές παραδέχονται ότι η Πολωνία είναι ένα κράτος μέλος όπου ο εισαγγελέας, οι εισαγγελικές αρχές θέλουν να μπουν στις λεπτομέρειες της υπόθεσης και να διευκρινίσουν τα ζητήματα. Κάποιοι κατηγορούμενοι και κάποιοι εκπρόσωποι ΜΚΟ είχαν υπογραμμίσει το θέμα της έλλειψης διαφάνειας, αλλά εδώ τα ζητήματα είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτό συμβαίνει. Ευχαριστώ. Ο κύριος ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να είναι η βασική αρχή επί των οποίων έχουν οικοδομηθεί οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Εγώ είμαι πολιτικός, έχω ζήσει υπό κομμουνιστικό απολυταρχικό καθεστώς και ξέρω σε τι βαθμό μπορούν να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ασφάλεια. Αυτά είναι τα βασικά δικαιώματά μας. Ξέρετε όμως ότι είχαμε τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Υόρκη, τον Παλί, τη Μαδρίτη, το Λονδίνο. Να μόνο μερικά παραδείγματα καταστάσεων όπου θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάστηκαν κατάφορα. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, όποιοι παραβιάζουν έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, δεν πρέπει να εκπλήσονται που δεν είμαστε πολύ τρυφεροί απέναντί τους. Χωρίς ε, έρευνες, ε, κανένας από τους εγκληματίες δεν θα μπορούσε να συλληφθεί. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τη στάση ορισμένου από τους συναδέλφους μας που επιτίθεται κατά των Αμερικανών συναδέλφων μας και ζητάνε από την Κομισιό να λάβει μέτρα. Όσο για τον κύριο Σνόντεν που κατηγορείται ότι παραβίασε το απόρριτο των πληροφοριών που γνώριζε το να προτείνεται το υποψήφιος για το βραβείο Ζαχάροφ είναι επίθεση κατά των αδέλφων μας. Ο κύριος Βόφς ένα λεπτό. Ευχαριστώ η τήρηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι στοιχείο κλειδί της πολιτικής της Ένωσης και γι' αυτό είναι προφανές ότι πρέπει να κάνουμε όλα όσα χρειάζονται για να τηρούνται αυτά τα δικαιώματα. Και πρέπει να ε, αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά τις παραβιάσεις τους. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε ποια προστιθεμένη αξία περιέχει αυτό το ψήφισμα που αύριο θα το ψηφίσουμε Έχουμε ψηφίσει για το θέμα αυτό το 2012 με βάση την έκθεση πρωτοβουλίας της ε, συναδέλφου Φλότρα η οποία ήταν ισορροπημένη, επί της ουσίας αποδεκτή και είναι σωστό βεβαίω να καλέσουμε το Συμβούλιο και την Κομισιόν να μας εξηγήσουν τι συνέχεια έδωσαν στο θέμα αυτό. Σωστό επίσης τα θέματα αυτά να τα επενθυμίζουμε, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν έχει έννοια και πάλι να αντιμετωπίζουμε το ίδιο περιεχόμενο και να επαναλαμβάνουμε αυτά που ήδη είπαμε και πέρυσι. Αυτό είναι ομφαλοσκόπηση. Γιατί το θέμα αυτό μπήκε στην ημερήσια διάταξη. Εφόσον έχουμε θέσει τα ερωτήματα. Επιπλέον το ψήφισμα βεβαίως ε, πηγαίνει και παραπέρα. Αυτά που αποφασίσαμε το 2012, πέρα από αυτά δηλαδή που πηγαίνει, που είχαμε αποφασίσει το 2012, και θέτει θέματα αρμοδιοτήτων αλλά και των δυνατοτήτων που έχουμε ως Ένωση. Πρέπει να ε, κινούμεθα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων μας. Πρέπει να βασιζόμαστε σε λογικές λύσεις και σας ευχαριστώ για την ε, προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόγκορ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. για λόγους ασφαλείας πρέπει να παίρνουμε τα αναγκαία μέτρα. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας χρειάζεται συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών. Των ε, μυστικών υπηρεσιών συμμάχων κρατών. Είναι απαραίτητη. Αυτό που διαπιστώνουμε εδώ είναι ότι εντός ευρωπαϊκών κρατών υπήρξαν πρακτικές που είναι σε απόλυτη αντίφαση προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία έχουμε οικοδομήσει εδώ και δεκαετίες και για τα οποία είμαστε περήφανοι. Εάν εμείς δεν παίρνουμε στα σοβαρά τους δικούς μας κανόνες, πώς θα καλούμε άλλους να πάρουν στα σοβαρά αυτούς τους κανόνες. Όλη αυτή η υπόθεση έχει συμβολική αξία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς επιπτώσεις, να μην τηρούνται διεθνείς συμφωνίες. Και μάλιστα ηθελημένα από κράτη-μέλη. Θέτουμε λοιπόν τη θεμελιώδη απέτηση, θέλουμε μια σαφή εικόνα για το θέμα αυτό για τον Ευρωπαίο πολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σόγκορ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα. Θέλετε να απαντήσετε κύριε Σόμπο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο Σόγκορ. Παρ' όλα αυτά ήθελα να ρωτήσω. Συμφωνούμε ότι η διερεύνηση αυτής της κατάστασης των φυλακών της CIA και άλλων παραβιάσεων των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι όλα αυτά θα πρέπει να είναι κυρίως αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων. Πρέπει να παίξουν μεγάλο ρόλο. Συμφωνώ κύριε Σόγκορ ότι η χώρα μας και η κυβέρνησή μας επίσης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην υπόθεση Σνόντεν. Και σε αυτά τα θέματα της CIA. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόγκορ. Ναι, μα είναι προφανές ότι συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι πρόκειται για αρμοδιότητα των κρατών μελών η διερεύνηση αυτών των υποθέσεων. Τώρα δεν θα αναφέρω όλα τα κράτη-μέλη που θα έπρεπε να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Δεν ξέρω τώρα να σας απαντήσω. Όσον αφορά τον κύριο Σνόντεν και τις φυλακές της CIA, όλα αυτά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Ένωση μπορεί βέβαια να βοηθήσει τα κράτη-μέλη αν δεν τα βγάζουν πέρα. Και τη Ρουμανία αφορά το θέμα αυτό. Εγώ είμαι από τη Ρουμανία. Δεν μπορώ να κάνω σχόλια για την Ουγγρική, ε, για την περίπτωση της Ουγγρατίας. Ευχαριστώ, κύριο Βαλέσα. 1,5 Ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Το σχέδιο ψηφίσματος περιέχει κάποια στοιχεία παράδεκτα κατά την άποψή μου. Οι κατηγορίες για έλλειψη διαφάνειας είναι ένα σημείο εγώ θέλω να τονίσω ότι οι δράσεις ε, των υπηρεσιών ασφάλειας αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή ε, εξελίσσεται ανεξάρτητη έρευνα στην Πολωνία που διεξάγεται από την ανεξάρτητη δικαστική αρχή. Η πολιτική πίεση λοιπόν που την κατεύθυνση αυτή είναι απαράδεκτη. Η έρευνα είναι υποεξέλιξη και το τελικό της από, η τελική της έκβαση θα εξαρτηθεί από την κρίση της εισαγγελία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο ζήτημα καθότι πολλά από τα έγγραφα βρίσκονται ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα. Τονίζω ότι η ασφάλεια των πολιτών μας αποτελεί το κύριο σημαντικότερο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η τρομοκρατία θέτει πάντα σε κίνδυνο τις αξίες μας. Αθώοι πολίτες της Ευρώπης γίνονται θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων από τρομοκρατικές ομάδες που χρησιμοποιούν διάφορα μέσα για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για την προστασία των πολιτών μας. Προφανώς σεβόμενοι το νομοθετικό πλαίσιο και διασφαλίσοντας ότι προσπίζουμε τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ο κύριος Λίσεκ, τελευταίος. Ευχαριστώ. Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, κυρίε και κύριοι, συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Γκόμες ότι πρέπει να αγωνιστούμε ενάντια σε αυτούς που παραβιάζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου και να μην δεχθούμε ποτέ να χρησιμοποιούνται παράνομες μέθοδοι κατά των φυλακιζόμενων. Αλλά υπάρχει κάτι που είναι άσχετο. Οι δηλώσεις, τα ανακοινωθέντα τύπου που περιλαμβάνουν κατηγορίες από φυλακισμένους ή ε, άτομα που έχουν συλληφθεί δεν μπορεί να είναι η βάση ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου. Εμείς σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν είχαμε τονίσει ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πολωνία μία ανακριτική δραστηριότητα. Θα συμφωνήσω με τους άλλους Πόλωνους συναδέλφους. Ο, η εισαγγελία της χώρας είναι η αρμόδια να κρίνει και τονίζω ότι η έρευνα βρίσκεται σε φάση στο τελικό της στάδιο και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να επιτρέψουν στις τοπικές αρχές να αναλαμβάνουν δράση σεβόμενη την αρχή της επικουρικότητας. Και κάτι ακόμα. Οι καταγγελίες αφορούν γεγονότα που έγιναν όταν στην κυβέρνηση ήταν η αριστερά. Ο κύριος Κβασνιεύσκη ήταν πρόεδρος ε, τότε, που αρνούνται το ότι υπήρξαν τέτοιες φυλακές. Τώρα φτάνουμε στη δικασία του ΚΑΤΣΔΙ. Ο κύριος Μέρφυ. Ευχαριστώ. Η Open Society Justice Initiative δημοσίευσε μία μελέτη που ε, επιβεβαιώνει αυτό που ήξερε η Ιρλανδία εδώ και χρόνια. Είναι μία από τις 15 ε, ε, χώρες που διευκόλυναν μέσω της παροχής εναέριου χώρου της επιχειρήσης της CIA στα πλαίσια αυτής της έκτατης έκδοσης, όπως ονομάζεται. Στο Σάνον υπήρχαν πολλά τέτοια αεροσκάφη. Βεβαίως, οι Αμερικανικές αρχές είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν θα μεταφέρονταν παρανόμως μέσα από την Ιρλανδική επικράτεια οι κρατούμενοι. Όμως είναι αναμφισβήτητο ότι όντως πέρασαν αυτές οι πτήσεις από την Ιρλανδία παραβιάζοντας έτσι τις διεθνείς συμβάσεις για τα βασανιστήρια. Όμως για να έχουμε αγαστές και ειδικέ εισαγωγικά σχέσεις με τη ΣΥΠΑ δέχθηκαν την κάλυψη, την απαγωγή και τα βασανιστήρια αυτών των κρατουμένων όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. τα μυστικά κέντρα κράτης πρέπει να κλείσουν, πρέπει να σταματήσουν αυτές οι πτήσει έκτατης έκδοση, πρέπει να απελευθερωθούν ή να απαγγελθούν επίσημες κατηγορίες αυτού του τους κρατούμενου, ώστε να έχουν μια δίκαιη δίκη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν βλέπω να υπάρχουν άλλοι ομιλητέ. Οπότε να καλέσω τον Υπουργό Λεσκεβίτσιου να πάρει το λόγο πλευρά του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της, ε, κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αξιότιμοι βουλευτές, το Συμβούλιο συμμερίζεται πλήρως την άποψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εθνούς δικαίου στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι θεμελιώδης. Διάφοροι ομιλητές σήμερα το απόγευμα κάλεσαν το Συμβούλιο να διερευνήσει ε, τους ισχυρισμούς ότι συμμετείχαν κράτη-μέλη σε ένα πρόγραμμα μεταφοράς και παράνομης κράτησης κρατουμένων από την CIA. Το Συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους των κυβερνήσεων των 28 κρατών μελών και ακόμη και αν είχε την νομική βάση να το πράξει το Συμβούλιο ποτέ δεν θα είχε πολιτική στήριξη από όλα τα 28 κράτη-μέλη για να κάνει μια δήλωση για τέτοια συμμετοχή πολύ λιγότερο να ξεκινήσει έρευνας. Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να είναι απογοητευτικό για τα μέλη του Κοινοβουλίου. Αλλά πρέπει να λειτουργούμε σε πλαίσια κανόνων που πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Αν υπάρχουν ισχυρισμοί απαράδεκτης συμμετοχής κρατών μελών σε τέτοιες δραστηριότητε, αυτό είναι πρώτα απ' όλα θέμα το οποίο πρέπει να διερευνήσουν τα εθνικά κοινοβούλια, οι εθνικές αρχές, εθνικές δικαστικές αρχές. Και υπάρχουν διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο για να τεθούν οι εθνικές κυβερνήσεις ενώπιον των ευθυνών τους. Βέβαια, μπορούν αυτές οι προσπάθειες να γίνουν και σε ευρύτερο επίπεδο, γιατί όλα τα κράτη-μέλη ε, συμμετέχουν και έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών. Υπάρχουν λοιπόν μηχανισμοί. Αλλά δεν είναι μηχανισμοί του οποίου ελέγχει το Συμβούλιο. Γι' αυτό το Συμβούλιο δεν έχει μπορέσει να δώσει συνέχεια στις συστάσεις που περιέχονται στο ψήφισμά σας. Δεν πρόκειται για έλλειψη διάθεσης ε, για ειλικρινή συνεργασία. Πρόκειται για θέματα νομικού και συνταγματικού πλαισίου εντός του οποίου πρέπει όλοι να λειτουργούμε. Γι' αυτό ε, παρακαλώ για την κατανόησή σας και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν σαφές. Έχουμε τέσσερις διαφορετικές προτάσεις. Θα ψηφίσουμε αύριο στις 12 από αυτόν. Λοιπόν, το επόμενο θέμα στην ημέρηση διάταξή μας είναι δήλωση της Επιτροπής και του Συμβουλίου για τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα λόγω των τραγικών γεγονότων στην Λαμπεντούζα. Πρώτος,